Αγαπητοί συνάδελφοι, πρωτού ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, μια σημαντική παρατήρηση, επιτρέψτε μου, την ε, Παρασκευή της εβδομάδας αυτής. Για τριακοστή φορά θα έχουμε την επέτειο της ε, συνθήκης ε, για την προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από 30 χρόνια αυτό σημαίνει ένα σημαντικό βήμα, γιατί δύο έθνη τα οποία επί σειρά δεκαετιών έζησαν δικτατορίας εντάχθηκαν στα, στη δημοκρατική κοινότητα λαών της Ευρώπης. 30 χρόνια αργότερα δεν μπορούμε να πούμε ότι τηρήσαμε κάθε δέσμευση και υπόσχεση, αλλά η δημοκρατία σίγουρα σταθεροποιήθηκε και ενισχύθηκε στις χώρες αυτές και η, ο αγώνας κατά των δικτατορικών δυνάμεων έχει σταθεί με επιτυχία. Σε αυτές τις ημέρες λοιπόν κυρίε και κύριοι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ισπανία και την Πορτογαλία, αντιμετωπίζουμε το εξής, οι υποσχέσεις που δίνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνοδευτεί και για, με την ευημερία για τους πολλούς, όχι για τον πλούτο για τους λίγους. Αυτό λοιπόν αμφισβητείται και φαίνεται και θα πρέπει να είναι κοινή βούληση όλων των πολιτικών δυνάμεων εδώ στο Κοινοβούλιο 30 χρόνια αργότερα να διασφαλίσουμε ότι αυτή η υπόσχευση για την ιστορική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική και οικονομική δύναμη της Ένωσης μετά τα, τις μεγάλες θυσίες που έκαναν οι λαοί της Ισπανίας και της Πορτογαλίας αυτή η υπόσχευση οικονομικής της δύναμης που οδηγεί σε ευμερία για τους πολλούς και για τις θέσεις απασχόλησης για τους νέους θα τηρηθούν αυτές οι υποσχέσεις από όλους από κοινό.